Θα ξεκινήσουμε λοιπόν συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε έχουμε την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα. Οργανώσαμε τη συνάντηση αυτή από κοινού με την αντιπροσωπεία για την Παλαιστίνη. Θέλω να καλωσορίσω λοιπόν όσους συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή των δύο οργάνων. Είναι μια συνάντηση η οποία χρονικά είναι ιδιαίτερος εύθετη θα έλεγα. Πιο πολύ από την τελευταία του μηνός Νοεμβρίου όταν με τον Πρόεδρο είχαμε συναποφασίσει να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα. Τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση στη Γάζα χειροτέρευσε έτσι περαιτέρω και όχι μόνο λόγω των περικοπών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για πάρα πολλούς άλλους λόγους, τους οποίους ε, είμαι βέβαιος ότι οι ε, ομιλητές μας θα παρουσιάσουν με επάρκεια. Από τις 30 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν οι λεγόμενες διαδηλώσεις της επιστροφής, Υπήρξαν πάρα πολλές συγκρούσεις την προηγούμενη Παρασκευή, για τέταρτη Παρασκευή, πυροβόλησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις με πάρα πολλά θύματα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 40 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών και εκατοντάλες άλλοι τραυματίστησαν και πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχασε και τη ζωή του ένα παιδί 15 ετών γιατί οι Ισραηλινοί στρατιώτες σημάδευαν στα κεφάλια των διαδηλωτών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 19 Απριλίου ένα κατεπήγον ψήφισμα Χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την κατάσταση λοιπόν στη Λωρίδα της Γάζας με αρκετούς εμπειρογνώμονες, τους οποίους έχει προσκαλέσει η Υποεπιτροπή με την Μανκούζη Ματέρη, εκπρόσωπη, εκπρόσωπο συγγνώμη, της Ούνρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Τζον Ντουγκάρντ, που είναι υπεύθυνο ε, ακαδημαϊκός για θέματα διεθνούς ποινικού από τις κάτω χώρες και τον Ασαλάμ υπεύθυνο ε, για μια οργάνωση που παρέχει ιατρική βοήθεια στους Παλαιστινίους και προσπαθεί να ενδυναμώσει το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Θα δώσω το λόγο απευθείας όμως για να μην καθυστερούμε στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη, τον κύριο Σιλικιώτη, για να κάνει και αυτός κάποιες λίγες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ το ε, καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Σέρφο Μπατζέρη. Να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση που διοργανώνουμε για αντιπροσωπεία σχέση με την Παλαιστίνη με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όντως η συνεδρία αυτή είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Όπω αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Μαντζέρη την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωκοινοβούλιο έκρινε κατεπίκο ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα τη Γάζα, σε συνέχεια τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τη ημέρα τη γη. Η ανθρωπότητα γίνεται για ακόμα μια φορά μάρτυρα του αληθινού προσώπου του Ισραήλ με τι Αναφορέ να είναι δραματικέ. Ε, από τι 29 του Μάρτη τουλάχιστον 45 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από πειράτων κατοχικών Ισραηλινών στρατικών δυνάμεων, ενώ οι τραυματίε είναι περίπου 2.000, εκ των οποίων οι περισσότεροι από του μισού από πραγματικά πειρά. Και 40 εξακολουθεί η κατάσταση να είναι κρίσιμη ε, στα νοσοκομεία. Όλα αυτά μαρτυρούν την αγριότητα και τη συστηματική καταστολή και καταπίεση της κρατική τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ σε βάρο των Παλαιστινίων. Συμπεριφορά του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινικά εδάφη καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του διεθνού δικαίου. Η χρήση βία και η σκόπιμη στοχοποίηση αμάθων συνιστά εγκληματική πράξη, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διεθνού έρευνα και οφείλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να συμβεί αυτό. Δηλαδή να υπάρξει μια διεθνής ανεξάρτητη επιτροπή για αυτά τα εγκλήματα. Πρέπει να σα πω ότι επειδή έγινε αναφορά και σε παιδιά, ε, μεταξύ αυτών έχασαν τη ζωή του και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο φορούσε διακριτικά πρέσ ε, και έπεσε από πειρά, μάλιστα βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από, το, από την, ε, τα σύνορα. Ε, οργή προκαλούν βεβαίω και οι, οι δολοφονίε τεσσάρων παιδιών την περασμένη εβδομάδα δολοφονήθηκε ο 15 χρονο Μουχάμετ Αγιούπ από πειρά Ισραηλινού στρατιώτη, μόνο ότι δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν, μάλιστα βρισκόταν σε μακρινή απόσταση. Ε, μέχρι σημείου τέτοιο αυτό το γεγονό που αναγκάστηκε ο ίδιο ο Ισραηλινό στρατό να ανακοινώσει ότι θα διαρρευνήσει έρευνα για το θάνατο του νεαρού Παλαιστινίου, ενώ η, Παλαι... η Παλαιστινιακή Αρχή ζητά από την ΟΗΑ ανεξάρτητη έρευνα για όλα τα επεισόδια στη Γάζα. Τα τραγικά αυτά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν την κλιμάκωση τη ένταση στη Γάζα και την αγανάκτηση ενό πληθυσμού που ζει συλλογικά φυλακισμένο περισσότερο από μια δεκαετία. Η Λωρίδα τη Γάζα, ένα μικρό κομμάτι τη γη, στο οποίο συνοστίζονται δύο εκατομμύρια άνθρωποι, βιώνει ένα ολοκληρωτικό αποκλεισμό από στεριά, θάλασσα και αέρα. Η Γάζα έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή φυλακή από τη βαβαρότητα του Ισραήλ. Οι κάτοικοι του στερούνται την ελευθερία αλλά και τα πιο βασικά ζωτικά αγαθά και υπηρεσίε, όπω την πρόσβαση σε νερό, σε διατροφή και σε υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ω αποτέλεσμα αυτού του 11χρονου απάνθρωπου αποκλεισμού έχουν αφήσει το 80% του πληθυσμού να εξαρτάται από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Και βεβαίω όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ουσιαστικό και αποφασιστικό ο ρόλο τη Ούντρα ε, για να μπορέσει να επιβιώνει αυτός ο πληθυσμός. Επιλέξαμε ακριβώς να εστιάσουμε τη συζήτηση στη Γάζα, γιατί είναι, εκεί είναι χειρότερη από οπουδήποτε αλλού στα κατεχόμενα την εδάφη. Και συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω των περιορισμών, έλλειψης ε, των βασικών αγαθών, όπως είπα προηγουμένως, της υγειονομικής περίστασης. Αυτή είναι η απελπισία του λαού που υποβάλλεται εδώ και μια δεκαετία σε ολοκληρωτικό ένα έργο χερσαίων και θαλάσσιων αποκλεισμών. Ε, να σας πω ότι σήμερα ε, θα ε, καλωσορίζουμε εδώ εμπειρογνώμενες. Αναφέρθηκε ο κύριος Παντζέρη, να αναφέρω και εγώ τους δύο που προσκαλέσαμε ως ε, αντιπροσωπεία της, του Ευρωκοινοβουλίου με Παλαιστίνη. Ο ένας καλωσορίζουμε εδώ το συνταγματάρχη Desmond Travers, ο Δέσμο Τράβη είναι μέλο τη ερευνητική αποστολή των ΕΕ για τη σύραξη στη Γάζα και ένα από του συντάκτε τη έκθεση Goldstone. Είναι απόστρατο συνταγματάρχη του Ιρλανδικού στρατού, ο οποίο υπηρέτησε σε διάφορε ειρηνευτικέ αποστολέ του ΟΗΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βασκάνια και τη Μέση Ανατολή. Σήμερα είναι αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Ποινικών Ερευνών. Το Ινστιτούτο Διεθνών Ποινικών ε, των Διεθνών Ποινικών Ερευνών προσφέρει κατάρτιση όσον αφορά τη διερεύνηση αποτροπαίων εγκλημάτων σε επαγγελματίε του τομέα τη ποινική δικαιοσύνη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, ε, ε, θα καλωσορίσω το Μαχμούτ Αμπου Ραχμάν, ο οποίο είναι Διευθυντή Επικοινωνίων και Διεθνών Σχέσεων στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αλ στη Γάζα, όπου διαμένει από το 2001 είναι κάτοχος μάστε στη θεωρία και πρακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο τη ΕΣΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου. Να σα πω ότι τον από Αμπουραχμά τον είχαμε πρόσφατα και σε συνεδρία τη αντιπροσωπεία με Παλαιστίνη, όπου συζητήσαμε για τι τελευταίε εξελίξει στη Γάζα την περασμένη Πέμπτη, τον οποίο και αυτό καλωσορίζω. Και ε, θα ξεκινήσω με τη συζήτησή μα ε, και θα δώσω πρώτα τον λόγο στην Έλενα Μασκούση Ματέρη, η οποία είναι Senior Liaison Officer of the UNRWA Representative Office στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο μας σε σένα, κυρία Ματέρη. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αντιπροσωπεία για σχέση με την Παλαιστίνη για την πρόσκληση που μας απευθύνεται θα ήθελα επίσης να εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική και οικονομική στήριξη προσφέρει στον οργανισμό μας, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ψήφισμα για την Γάζα και γι' αυτό είμαστε επίσης ευγνώμονες. Μετά από τις παρεμβάσεις των δύο συμπροέδρων, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τα πρόσφατα επεισόδια στην Γάζα στη διάρκεια διαδηλώσεων που γίνονται ήδη από την 30η ε, Μαρτίου. Τρεις σπουδαστές έχασαν τις ζωές τους σήμερα και άνω των 100 αναφέρονται ότι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές. Με την ευκαιρία ωστόσο θα ήθελα να σας αναφέρω και για τα σοβαρά προβλήματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουμε στην Γάζα και ιδίω για Παλαιστίνιους πρόσφυγες άνω του 1,5 εκατομμυρίου στην ε, Λόριδα της Γάζας. Έχουμε εντολή να παρέχουμε υποστήριξη σε 5 εκατομμύρια Παλαιστινίους Λωρίδα της Γάζας, Ανατολική Ιερουσαλήμ κλπ. με τις δραστηριότητές μας που αναφέρονται σε υγεία, παιδεία, άλλες υπηρεσίες, μακροοικονομική στήριξη, καθώς και βοήθεια για κατεπίγουσες καταστάσεις. Πράγματα τα οποία συμβάλλουν στην ε, ανόρθωση των δικαιωμάτων εκπαίδευσης. Παρακαλείτε ομιλείτε αν μπορεί να διαβάζει λίγο πιο αργά. Λίγο πιο αργά θα μας διευκολύνει όλα αυτά στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες είναι σε μια κατάσταση που χαίρουν προστασίας για το μακρότερο χρονικό διάστημα. 5,3 εκατομμύρια ή 23% του συνολικού ε, προσφυγικού πληθυσμού ανά τον κόσμο. Τον επόμενο μήνα θα είναι η 70η επέτειος από, την, από τον αρχικό τους εκτοπισμό, δηλαδή τρίτη γενιά Παλαιστινίων που ζουν χωρίς δίκαιη επιστροφή στα εδάφη τους. Πολλοί έχουν υποστεί σοβαρότατα τραύματα από τους διάφορους διαδοχικούς κύκλους βίας ήδη από το 1949. Και αυτό ισχύει ιδίω για αυτούς που διαμένουν στη λωρίδα της Γάζας, που ε, σε αυτήν βρίσκονται 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι ο αποκλεισμό της λωρίδα της Γάζας μπαίνει στο 10ο χρόνο του τον Ιούνιο. Τα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη να αρθεί ο αποκλεισμό και να απαγορευτεί, ούτως ή άλλως απαγορεύεται υπό το ε, διεθνές δίκαιο ως συλλογική τιμώρηση. Πρέπει να αποκατασταθεί το δικαίωμα της ελευθερίας διακίνησης καθώς και τα πολιτιστικά τους και πολιτικά τους δικαιώματα και να ανυψωθεί το βιωτικό τους επίπεδο. Μικρός αριθμός ανθρώπων λαμβάνουν άδειε εξόδου, μεταξύ αυτών επιχειρηματίες. Ο αριθμός ασθενών που ζητούν άδεια για να εξέλθουν από τη πλευρά της Γάζας έχει διπλασιαστεί από το 2012, αλλά ο ρυθμός των εγκρίσεων από τις ε, Ισραηλινές αρχές μειώνεται από 92% το 2012 σε 62% το 2016 και 55% τον Οκτώβριο του 2017. Η ελευθερία της διακίνησης παρεμποδίζεται επίσης και προς την Αίγυπτο. Στους πρώτους δύο μήνες τούτου του χρόνου, του 2018, το άνοιγμα της Ράζα άνοιχτηκε εν μέρη από τις Αιγυπτιακές Αρχές μόνο για 7 ημέρες. Φέτος μόνο για 36 ημέρες. Πράγματι, οι περισσότεροι από αυτούς που διαμένουν στη Γάζα δεν μπορούν να φτάσουν στον έξω κόσμο, ούτε βεβαίως και στα λοιπά κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Έχουν λοιπόν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στον κόσμο, 43% σε ό,τι αφορά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δε είναι 75% και για τις γυναίκες 66%. Εμείς είμαστε οι δεύτεροι μεγαλύτεροι εργοδότες μετά από τις δημόσιες αρχές και για την παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα. Εκτός από αυτό, κάνουμε προσπάθεια να ελαφρύνουμε την πίεση στις ε, παλαιστινιακές οικογένειες, δίνοντας δυνατότητες σε σύντομη έστω απασχόληση σε μέλη τους. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά άνω του 80% του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Και μετά από το 2016 η πιο σημαντική ανθρωπιστική παρέμβαση είναι η παροχή τροφίμων. Η διατροφική ασφάλεια έχει επιδεχθεί σημαντικά. Ο αριθμός των Παλαιστινίων προσφύγων από 80.000 το 2000 έχουν φτάσει σήμερα το 1 εκατομμύριο που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική παροχή τροφίμων με σημαντικές ε, επιπτώσεις στην υγεία τους. Έχουμε κάνει μελέτη με 2.000 πρόσφυγες και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάνω από το μισό δείγμα των προσφύγων τις κάνουν πάλι νόημα να μιλεί πιο αργά, ε, αν είναι δυνατόν να μιλήσει λίγο πιο αργά. Μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπίζουν επίση βαρύτατε δυσχέρειε από την άποψη αυτή. Ιδίω η νεολαία θίγεται μεταξύ τη υψηλή ανεργίας και κάποιων ειδών απασχόλησης που είναι απολύτω ε, ανεπαρκείς και αβέβαιε. Το αποτέλεσμα είναι μία αίσθηση του κόσμου ότι δεν αποδίδουν οι επενδύσεις στην παιδεία και μια βαθιά απογοήτευση διότι δεν υπάρχει καμιά πολιτική πρόοδος, μια πολιτική λύση. Η Άννα απευθύνει έκκληση προ όλου. Η συλλογική μα ευθύνη είναι να αποδείξουμε ότι δεν έχουν δίκιο στην αίσθηση αυτή. Από τα πιο πιεστικά θέματα σήμερα είναι η μεγάλη έλλειψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματο. Το 2012 με μια μελέτη είχαμε δει ότι το 2020 θα είναι πλέον ακατοίκητη η λωρίδα της Γάζας. Εξακολουθεί η παρακμή αυτή από κάθε άποψη. Για το ηλεκτρικό ρεύμα έχει χρόνια έλλειψη η Γάζα. Από το 2017 στα μέσα του χρόνου σημειώθηκε σοβαρή μείωση και πολλοί Παλαιστίνοι στην Γάζα δεν είχαν παρά μόνο 4 ώρες ηλεκτρικό ρεύμα το 24ωρο. Η κατάσταση του νερού είναι ακόμα πιο οξία. Γνωρίζουμε ότι 1,2 εκατομμύρια των κατοίκων της Γάζας δεν έχουν ε, τρεχόμενο νερό. Αυτό επιδεινώνει την κατάσταση ιδίως των προσφύγων και ακόμα περισσότερο των παιδιών. Πολλοί από τους οποίους ε, ε βρίσκονται σε κίνδυνο να κολλήσουν σοβαρές ασθένειες που οι παθογόνοι οργανισμοί τους μεταφέρονται με τα απόβλητα και δεν επιτρέπει στους κατοίκους της Γάζα να ζήσουν φυσιολογικά τη ζωή τους. Η Ούνρα ζητά λογοδοσία. για τα όσα έγιναν με τις θεοπραξίες του 2013 και ζητούμε και επίσης βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων εκείνων των επεισοδίων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων της Γάζας δεν μπορεί να διαχωριστεί από την οικονομική κατάσταση και των οργανισμών μας. Η Άνρα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική χρηματοδοτική κρίση με την απόσυρση σημαντικού τμήματος χρηματοδότησης από το πιο σημαντικό της δωρητή φέτος, χωρίς δηλαδή τον ομφάλιο λόρο που χρειάζεται η Γάζα για να προσφέρει, η Ούρα δηλαδή, για να προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας. Και παιδεία για 270.000 σπουδαστές στη Γάζα, οι οποίοι πηγαίνουν καθημερινά στη σχολεία της Άνδρα. Για εγγύους γυναίκες, για παιδιά και για ηλικιωμένους που όλοι αυτοί εξαρτώνται από τις δικές μας προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας των προσώπων αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διαφυλαχθούν. Ο πληθυσμό τη Γάζα, ιδίω εν ώψη των πρόσφατων επεισοδίων, αρχίζει και διαρωτάται αν εφαρμόζεται πράγματι το διεθνέ δίκαιο στην κατάστασή του. Για άλλη μια φορά η Άνδρα ζητεί ε, ανάληψη συλλογική ευθύνη και αποφασιστικότητα από τη διεθνή κοινότητα για να αποδείξουμε στα πρόσωπα αυτά ότι εν τέλει έχουν άδικο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ματέρη τώρα το λόγο έχει ο Professor John Dukart, το former Special Rapporteur of the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory. The floor is yours, Professor. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι γεγονός ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, έχουν διαπραχθεί στη Γάζα. Στα πλαίσια των τελευταίων παρεμβάσεων του Ισραήλ και στα πλαίσια επίσης και των τελευταίων διαμαρτυριών των Παλαιστινίων. Μετά την επιχείρηση του 2009 ήμουν υπεύθυνο της αντιπροσωπείας που πήγε για να ελέγξει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και ε, διαπιστώσαμε την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Έχει αποκλειστεί και είναι παράνομο αυτό φυσικά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά. Είναι επίσης δεδομένο ότι το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά και σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να πούμε ότι τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή κυβέρνηση υπέβαλε μία αναφορά στα πλαίσια των διαμαρτυριών για την διακρίσεις, τις φιλετικές, γιατί το Ισραήλ ουσιαστικά ασκεί ένα απαρτχάιντ στην ε, Λωρίδα της Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Είναι πρώτη φορά που κατατίθεται μια τέτοια αναφορά στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης και έχουν πλέον το θάρρος για να καταθέσουν την διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος μεταχειρίζεται τους πολίτες του. Βασίζεται λοιπόν η καταγγελία στις φιλετικές διακρίσεις και ζητά την δημιουργία μιας ειρηνευτικής επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο θα έχει νομίζω συνέπειες πολιτικές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τους διεθνείς μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική απόδοση ευθυνών στην ε, περιοχή αυτή. Συνάντησα έναν δανό διπλωμάτη όταν ήμουνα στη Γάζα, ως ειδικό εισηγητής ε, για την κατάσταση, στα κατεχόμενα. Ο δανός αυτός διπλωμάτης ερευνούσε τις ζημίες που είχαν προκληθεί σε ένα σχέδιο, σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε η Δανία, ένα σχολείο μάλιστα, το οποίο το Ισραήλ το κατέστρεψε πάρα πολύ απλά και συνέλεγε ο Δανός διπλωμάτης πληροφορίες ε, για την καταστροφή αυτή και προσπαθούσε να αξιολογήσει την καταστροφή. και θεώρησε ότι θα έπρεπε να ζητηθεί, τον, τον ρώτησα μάλλον, αν θα α, υπάρξει αίτημα για αποζημίωση από το Ισραήλ και μου είπε ότι καλά τώρα αυτά είναι αστεία. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει το θάρρος να ζητήσει τέτοια πράγματα από το Ισραήλ. Οι, οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία κάνει το Ισραήλ είναι λάθος, γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία κάνει το Ισραήλ είναι παράνομα, γνωρίζουν ότι έχουν διεθνείς μηχανισμούς για την λογοδοσία στο Ισραήλ, αλλά αποφασίζουν να μην κάνουν τίποτα. Τώρα να αναφερθώ λίγο στους βασικούς διεθνείς μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Καταρχάς υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ποινικό δικαστήριο, υπεύθυνο για, για θέματα ποινικά σε διεθνές επίπεδο, για εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Η Παλαιστίνη είναι κράτος μέλος, στο έδαφος της έχουν διαπραχθεί εγκλήματα στην Ιερουσαλήμ, στην Δυτική Όχθη, στην Γάζα. Αλλά φυσικά το Ισραήλ έχει αποφασίσει για ευνόητους λόγους να μην ε, είναι τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου έχει ξεκινήσει από το δικαστήριο μία προκαταρτική μελέτη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία διεπράχθησαν στα Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου του 2015 η προκαταρτική έρευνα και συνεχίζεται. Στόχος είναι να αποφασιστεί αν υπάρχουν βάσιμες υποψίες έτσι ώστε να ασκηθούν διώξεις. Αυτή η προκατακτική έρευνα συνεχίζεται τώρα για 3,5 χρόνια. Το θέμα αυτό ήταν προς εξέταση από το Διεθνές Ποινικό 9 χρόνια. Ήδη από το 2009 και μετά από τις δολοφονίες που είχαν διαπραχθεί ε, εις βάρος ε, της ε, ανθρωπιστικής αποστολής Μαβή Μαρμαρά. Υπάρχουν και άλλα διαβήματα τα οποία έχει ξεκινήσει η Παλαιστινιακή Κυβέρνηση και Παλαιστινιακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η εισαγγελία του Διεθνούς Δικαστηρίου ε, έχει πλέον στοιχεία στη διάθεσή της, αλλά είναι σαφές ότι ασκούνται πιέσεις, κυρίως από το Ισραήλ και τις Ηνωμένε Πολιτείες και είναι ε, ανοιχτό πια μυστικό ε, το ότι τα ευρωπαϊκά κράτη είναι αντίθετα με την ιδέα δίωξης του κράτους του Ισραήλ και πιέζουν έτσι ώστε να μην αναλυθεί δράση εις βάρος του. Η σύσταση την οποία δίδω εγώ είναι ότι αν τα κράτη-μέλη θέλουν να αποφύγουν κατηγορίες ότι είναι συνένοχοι στην αποτυχία της εισαγγελία να δώσει συνέχεια στη δίωξη, να διευκρινίσουν ότι θα στηρίξουν τις ενέργειες της εισαγγελία και σε δημόσιο επίπεδο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο έτσι ώστε να αποκτήσει ο εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού το φάρος αν θέλετε και την όρμη να προχωρήσει στην άσκηση δίωξης εις βάρος του Ισραηλινού κράτους. Αυτός είναι ο πρώτος μηχανισμός. Ο δεύτερος μηχανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ο διακρατικός μηχανισμός για φυλατικές διακρίσεις. Ξέρετε όπως σας είπα ότι η Παλαιστίνη ξεκίνησε με μία αναφορά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργάνωση να στηρίξει την αναφορά την Παλαιστινιακή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Ή και να καταθέσουν και οι ίδιες αυτές οι χώρες αντίστοιχες αναφορές για την καταγγελία του Απαρτχάιντ στα κατεχόμενα. Ένα τρίτο μέσο είναι η λεγόμενη διεθνής δικαιοδοσία εθνικών δικαστηρίων. Αυτό επιτρέπει σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να στραφεί εναντίον ενός ας πούμε αξιωματικού Ισραηλινού ή ενός πολιτικού Ισραηλινού λόγω διάπραξης πολιτικών εγκλημάτων. Είναι μια αρχή καθιερωμένη ε, στο διεθνές δίκαιο τα τελευταία χρόνια όμως τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αρχίσει και βάζουν τροχοπέδι στη, στην πρακτική αυτή. Ελπίζω να ξεκαθαριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να επιτρέπουν την λεγόμενη καθολικού τύπου δικαιοδοσία σε εθνικά δικαστήρια. Και τέταρτο μέσο και τελικά και επανέρχομαι στον δανό διπλωμάτη της αρχής της παρουσίασής μου, θα πρέπει να ενθαρρυθούν τα κράτη-μέλη να ζητήσουν αποζημίωση από το Ισραήλ για τις ζημίες ε, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ε, και υποδομών στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, κυρίως στη Γάζα. Κλείνοντας θα πρέπει να πω το εξής και νομίζω ότι έχει σημασία. Τα κράτη-μέλη διστάζουν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και να εξαναγκάσουν το Ισραήλ. Δεν θέλουν καταρχάς να σταθούν αντίθετοι στην Αμερικανική πολιτική. Δεύτερον, επηρεάζονται από τα Ισραηλινά λόμπι. Τρίτον, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τις λεγόμενες τύψεις του ολοκαυτώματος. Και τέταρτον, Οι πολιτικοί σε ορισμένες χώρες δεν θέλουν να καταγγέλουν το Ισραήλ γιατί φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν για αντισημιτισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε λίγο να διευκρινιστεί ότι αντισημιτισμός δεν σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση μίσος εναντίον των Εβραίων, αλλά ε, καταγγελία σαφής και ξεκάθαρη για τις ενέργειες του Ισραηλινού κράτους τα κατεχόμενα εδάφη. Η προσπάθεια που κάνει το Ισραήλ να διευρύνει την έννοια του όρου αντισημιτισμός είναι ένα εμπόδιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ ασκεί apartheid στα Παλαιστινιακά εδάφη. Δεν ξέρω αν είναι του ιδίου τύπου με αυτό της ε, Νοτιού Αφρικής ή χειρότερο. Θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι Νοτιοαφρικανοί οι οποίοι έχουν πάει στην Παλαιστίνη θεωρούν ότι είναι χειρότερη μορφή apartheid αυτή που ασκείται εκεί από ό,τι στη Νότια Αφρική. Έχει σημασία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να είναι πιο θαραλέα απέναντι στο Ισραήλ αν δεν το κάνει αυτό, ε, δίκαια θα κατηγοριστεί για συνενοχή σε εγκλήματα τα οποία διαπράττει η χώρα του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Thank you, Professor John Dugart. Uh, and now I give the floor to Dr. Δίνω το λόγο τώρα στον δόκτωρα Καλύτερα να ακούσουμε πρώτα όλες τις τοποθετήσεις και μετά. Και μετά ερωτήσεις. Ιατρικό σύμβουλος. Η ιατρική, η medical aid δηλαδή για την ε, Παλαιστίνη. Ε, αυτό που κάνουμε είναι να προσφέρουμε ιατρική βοήθεια. Έχουμε γραφεία στον Λίβανο, εκεί ε, άλλωστε κάνουμε ε, τα ίδια και στην Γάζα. Σήμερα θα ρίξω το φως ιδίως στην Γάζα. Έχουμε τρεις τομείς, emergency, μητρική βοήθεια σε μητέρες δηλαδή, πρωταρχική βοήθεια σε παιδιά, ανθρώπους με αναπηρίες και ψυχολογική στήριξη. Έφυγε το Ισραήλ το 2005 από, το, από τη Γάζα, αλλά διατηρεί έλεγχο στον πληθυσμό και ως ε, δύναμη κατοχής έχει όλη την ευθύνη και για τα ανθρωπιστικά, όπως προκύπτει από την τέταρτη συνθήκη της ε, Γενέβης και από τα σχετικά με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Το αποτέλεσμα του αποκλεισμού της Γάζας όμως έχει καταστρο... καταστρεπτικές συνέπειες στην οικονομία της Γάζας και οδήγησε επίσης και στην ε, ε, διάλυση του τομέα υγείας. Περιορισμοί για την έξοδο των επαγγελματιών υγείας από τη Γάζα τους, ε, δεν τους επιτρέπει να εκπαιδεύονται. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών σε πολλούς τομείς όπως ε, χειρουργική, οφθαλμιατρική κλπ. Και επίσης ο περιορισμός των ε, εισαγωγών λεγόμενων δυτής χρήσης ε, μηχανημάτων δεν επιτρέπει την εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων και ακόμη και ηλεκτρικών εργαλείων που χρειάζονται για την λειτουργία τους. Επίσης τα αναλώσιμα αγαθά βρίσκονται σε μεγάλη έλλειψη το Φεβρουάριο του 2018 και πριν να αρχίσουν οι πολλές απώλειες. 23% αναλωσίμων, ειδών αναλωσίμων δηλαδή, δεν έχουν επαρκή αποθέματα. Εξάλλου, έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που ε, κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη λειτουργία των νοσοκομείων. Η λειτουργία τους περιορίζεται σε 4-5 ώρες. Ε, το δε καύσιμο για τις γεννήτριες που υποτίθεται ότι θα δίνουν ρεύμα σε περιπτώσεις διακοπής, ε, πάλι ε, είναι πανάκριβο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι σημαντικό οι ασθενείς να μπορούν να μεταφέρονται εκτός της Γάζας για να λαμβάνουν τη θεραπεία που δεν μπορεί να τους προσφερθεί εντός του κατεχόμενου δάφους της, εντός μάλλον της Λωρίδας της Γάζας. 54% όμως των εγκρίσεων για το 2017 και σκεφτείτε ότι το 2012 οι εγκρίσεις ήταν 92% εγκρίσεις εξόδου. Πέραν αυτού, η φροντίδα υγείας έχει αντιμετωπίσει πολλές επιθέσεις και το 2009 και το 2012 και το 2014. Στην επίθεση εκείνη, 73 νοσοκομεία και κλινικές υπέστησαν ζημίες και καταστράφηκαν. Και καταστράφηκε ολοσχερός και το μόνο νοσοκομείο αποκατάσταση. 45 νοσοκομιακά αυτοκίνητα καταστράφηκαν και 78 ε, νοσηλευτές ή ιατρικό προσωπικό ε, τραυματίστηκαν και ένα αριθμό σκοτώθηκε. Τα, οι επιπτώσει αυτέ δεν είναι μόνο άμεσες σε ό,τι αφορά δηλαδή, την καταστροφή αλλά και τις απόλυσεις ανθρώπινων ζώων. Δεν επιτρέπει και την προσφορά φροντίδων υγεία, μακροπρόθεσμα. Η δε ατιμορρησία για επιθέσει κατά ιατρικών, ιατρικού προσωπικού και κλινικών νοσοκομείων κλπ. δημιουργεί ένα κλίμα που επιτρέπει βαρύτατες ε, παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και από το 2014 η οργάνωση Medical Aid for Palestinians συνεργάζεται με τους εταίρους μας στέλνοντας ορθοπαιδικούς χειρούργους από το King's College στο Λονδίνο για να κάνουν εγχειρήσεις σε, σε ε, ασθενείς και επίση να έχουν στήσει και ένα εργαστήριο εκεί για να φτιάχνουν τεχνητά μέλη και εκπαιδεύουν γιατρού και νοσηλεύτριες. Και το 2015 με αυτό το κέντρο στο νοσοκομείο ΣΕΦΑ. Έργο το οποίο ήταν ζωτικό για να ανταποκριθούμε στις ε, τρέχουσες ε, περιστάσεις. Οι απαντήσεις του Ισραήλ τώρα στις διαδηλώσεις από την 30η Μαρτίου ήταν πολύ βίες από την 30 Απριλίου μέχρι προχθές έχουν πάνω από 1240 τραυματισμούς. Μάλλον 1539 από πυροβολισμούς, πολλές εκατοντάδες από εισπνοή αερίων και τέλος και από χρήση ελαστικών σφαιρών. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις των διεθνών οργανώσεων δείχνουν 37 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες. 3.268 κατέληξαν στα νοσοκομεία και πιστεύουμε ότι αν συνεχίσει ο ρυθμός αυτός από πολιών θα φτάσουν πάνω από 7.600 νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία. 70% δηλαδή του αριθμού που είχαν ε, τραυματιστεί στην επίθεση στη Γάζα του 2014. 17% από όλα αυτά τα θύματα είναι παιδιά. 20 ασθενείς ζήτησαν να εξέλθουν από τη Γάζα για να λάβουν ε, θεραπεία. 9 μόνο έγιναν δεχτές, δηλαδή 45% και 15% από το συνολικό 65% για το πρώτο τρίμηνο του 2018 και ε, στις 11 αρνήθηκαν. 55% βεβαίω είναι υψηλότερο από το 8% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και από την 30 Μαρτίου μέχρι την 23η Απριλίου τουλάχιστον 77 νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό τραυματίστηκαν και 14 νοσοκομιακά αυτοκίνητα καταστράφηκαν σύμφωνα με τον οργανισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μισελίνου. Κυρίως πρόκειται για τραυματισμούς των κάτω άκρων με καταστροφή ή γονάτων από, ή, ε, των κάτω ε, άκρων από ε, σφαίρες. Τουλάχιστον 17 ακροτηριασμοί έχουν καταγραφεί ως τώρα, 4 στα άνω άκρα και 13 στα κάτω και αναμένονται και άλλοι. Θα σας διαβάσω τώρα μία δήλωση από ένα γιατρό επιτόπου στη Γάζα. Οι σφαίρες που χρησιμοποιούν προκαλούν τραυματισμούς που δεν έχουμε ξαναδεί από το 2014. Ενώ η είσοδος της σφαίρας είναι μικρή, η οποία εισόδου δηλαδή, η οποία εξόδου είναι τεράστια. Και χρειάζονται και ορθοπαιδικό και πλαστικό χειρουργό για να διασώσουν τα άκρα αυτά. Η Γάζα δεν έχει τέτοιε δυνατότητε. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν τραυματίε με, βαριές, με, βαριές, με βαριά τραύματα τα οποία μολύνονται. Και μόλι πάμε κάπω να πάρουμε ανάσα, έρχεται νέο κύμα τραυματιών από την επόμενη Παρασκευή. Πράγματα τα οποία δεν θα άντεχαν ούτε τα καλύτερα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Φανταστείτε τώρα νοσοκομείο στη Γάζα με τι ελλείψει που αντιμετωπίζει και σε προσωπικό και σε αναλώσιμο και Και αυτά συμβαίνουν κάθε Παρασκευή. Έχουμε κάνει έργο αποκατάστασης εδώ και χρόνια και τα αποτελέσματα είναι ε, αυτή τη στιγμή διακυβεύονται. Η οργάνωση Medical Aid for Palestinians ανησυχεί επίσης και από τη χρήση ε, μη θανάσιμων όπλων. Αυτά που λέγονται control devices, δηλαδή πλαστικές ή λαστιχένιες σφαίρες επίσης δακρυγόνα, τα οποία επίσης μπορούν να προκαλέσουν βαριούς τραυματισμούς ή και θάνατο και κυρίως αν βληθούν από ε, μικρή απόσταση ή αν κτυπήσουν το θύμα ας πούμε στο στήθος ή στο κεφάλι. Και τώρα θα σας πω για μια περίπτωση που βρήκαν οι γιατροί που έμειναν πραγματικά αμήχανοι όταν ε, έκαναν την εγχείρηση αφαίρεσαν από το κεφάλι ενός ε, ασθενούς, ενός τραυματία δηλαδή, ε, μικρό σακί με μολυβένιους βόλους που είχε μπει 5%, ε, 5 εκατοστά μέσα στο κρανίο του ανθρώπου αυτού. Μετά από 4 ώρες χειρουργείο ο άνθρωπος αυτός ζούσε ακόμα. Τέτοιου είδους βλήματα δεν είναι βλήματα ακριβίας και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Και πολλά τέτοια βλήματα κτυπούν το σώμα του θύματος με πάρα πολύ μεγάλη ορμή και προκαλούν βαρύτατους τραυματισμούς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εργαζόμαστε και η ανταπόκριση που δίνουμε μαζί με την ICRC και τους ιατρούς χωρίς σύνορα είμαστε από τους πρώτους που τρέχουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όλες οι αποκαταστάσεις άκρων που κάνουμε και οι ε, γιατροί μας ξεκίνησαν τις 30 Μαρτίου με υλικό το οποίο κοστίζει 130.000 δολάρια και το οποίο καταναλώθηκε μέσα σε 24 ώρες. Ε, στέλνουμε και αναλώσιμα, στέλνουμε και ε, σακούλες με αίμα και συνεχίζουμε να στέλνουμε τέτοια υλικά. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συλλέξουμε ένα εκατομμύριο δολάρια για να μπορέσουμε να στείλουμε περισσότερα φάρμακα και αναλώσιμα καθώς και άλλα υλικά και στέλνουμε και ορθοπαιδικό χειρουργό σύμβουλο για 10 ημέρες στην Γάζα για να υποστηρίξει τα πρόσωπα που κάνουν ε, τις επιχειρήσεις και ελπίζουμε θα μπορέσουμε να στείλουμε και ειδικό για ανάπλαση ε, αιμοφόρων αγίων. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προστατευτούν σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, που σημαίνει ότι χρειάζεται ανεξάρτητες έρευνες για να δουν εάν χρησιμοποιούνται όπλα ελευθέρων σκοπευτών και άλλα τα οποία κατασκευάζονται στο Ισραήλ και αν χρησιμοποιούνται για την παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χρειάζεται επίσης προστασία το ιατρικό προσωπικό και εγκαταστάσεις Ελπίζουμε ότι οι χώρες μέλη θα ανταποκριθούν στις ανάγκες άμεσης προστασίας και παροχής ιατρικών ομάδων για αντιμετώπιση κατεπιγουσών περιπτώσεων, καθώς επίσης και με την παροχή αναλώσιμων φαρμάκων κλπ. Αλλά πρέπει να γίνει μια ε, σοβαρή επένδυση μακροπρόθεσμα για παροχή υγείας, φροντίδων υγεία δηλαδή, στον Παλαιστινιακό πληθυσμό παρόλο τον, παρόλο τον Ισραηλινό αποκλεισμό και βεβαίως την Ισραηλινή στρατιωτική κατοχή. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Desmond Travers. μέλος της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής Διερεύνησης της κατάστασης στην Παλαιστίνη, στα κατεχόμενα εδάφη. Θα ήθελα να βασιστώ στην, στο PowerPoint το οποίο έχω ετοιμάσει. Θα αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην διάμεση περιοχή ανάμεσα στη Γάζα και στο Ισραήλ. το θέμα των πυρομαχικών, των μη κατάλληλων πυρομαχικών είναι ένα σοβαρό θέμα και θα ήθελα στο τέλος παρουσίασής μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις γύρω από αυτό. Αυτά τα οποία συνέβησαν στην ενδιάμεση ζώνη, στη διαχωριστική ε, περιοχή δεν είναι πρόσφατα μόνο βασίζονται στην στρατιωτική αποστολή της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και 21ης Ιανουαρίου του 2009 των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας. Στα πλαίσια αυτής της αποστολής υπήρχε και μία επιπλέον αποστολή από πλευράς του μηχανικού του στρατού. Έφεραν μπουλντόζες και ε, καθάρισαν την περιοχή ε, για 1500 τετραγωνικά μέτρα, καταστρέφοντας ε, εκριζώνοντας χιλιάδες ελαιόδένδρα, χιλιάδες δέντρα με σπεριδοειδή και καταστρέφοντας ολόκληρες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό δημιούργησε κατ' ως στρατιωτικό. όχι μια ζώνη προστασίας, αλλά μια ζώνη ελευθέρων σκοπευτών. Το λέγω αυτό. Γιατί από το τέλος της αποστολής αυτής, όταν αμφισβητήθηκε η συμπεριφορά των Ισραηλών, that Israeli military would contain... Οι συμπεριφορές αυτές ε, στην αρχή δεν είχαν γίνει ιδιαίτερα κατανοητές. Οι στατιστικές δείχνουν ότι για τα επόμενα τρία χρόνια αυτή η ζώνη προστασίας ε, ε, μετετράπει όπως είχαμε προβλέψει τότε σε μια ζώνη θα έλεγα ελευθέρων σκοπευτών. Συνεπώς η αποστολή του 2009 η επιχείρηση του 2009 ήταν στρατηγική επιχείρηση και σε συνεργασία με ε, την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της ζώνης, της ενδιάμεσης, της ζώνης προστασίας, ε, δημιουργήθηκαν και άλλα προηγούμενα αρνητικά για τη Γάζα. Κατέστρεψαν σαν παράδειγμα τον τελευταίο αλευρόμιλο εισάγεται πλέον το αλεύρι, οπότε υπήρξε θέμα έτσι κι αλλιώς σε σχέση με τα τρόφιμα. Κατέστρεψαν επίσης με πολύ συγκεκριμένο και στρατηγικό τρόπο την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Και φυσικά αυτό δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα μόλυνσης των του υδάτινου ε, ορίζοντα, ο οποίος τώρα πλέον είναι ιδιαίτερα μολυσμένος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και φυσικά αυτό ε, μόλυνε και τα παράκτια ύδατα. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα ε, κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής της επιχείρησης του 2009 που αποδεικνύουν ότι υπήρχε στρατηγική προσπάθεια καταστροφής των στρατηγικών λειτουργιών της Γάζα. Η αστυνομία, σαν παράδειγμα, ήταν πολύ αποτελεσματική. Είχε αντιμετωπίσει τις τοπικές μαφίες και τα στοιχεία τα εγκληματικά. Ε, στοχεύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε μία επίθεση μάλιστα το 2009 όταν έκαναν παρέλαση οι αστυνομικοί της Γάζα ε, στην ουσία δολοφονήθηκαν 88 αστυνομικοί λέει ο μιλητής. Οικονομικά λοιπόν η προσπάθεια αυτή ήταν ε, καταστροφική. Στην ουσία ε, ενσωματώθηκε σε αυτή την νεκρή ζώνη το 68% του καλλιεργούμενου εδάφους, του αρρώσιμου εδάφους ε, της ε, περιοχής αυτής της Γάζα. Οι εξηγήσει τις οποίες ε, δίδει το Ισραήλ είναι ότι στην ουσία ήταν αυτάρκης η λωρίδα της Γάζα και γι' αυτό δεν υπήρχε πρόβλημα με την καταστροφή αυτής της μεγάλης έκτασης. Μετά υπήρξε και η αποστολή Protective Edge, η επιχείρηση Protective Edge. Χρησιμοποιήθηκαν τεράστιες ποσότητες ε, πολεμοφοδίων. Από τον αέρα, από το έδαφος, χιλιάδες τόνοι πυρομαχικών έπεσαν στη λωρίδα της Γάζα. Αυτό το οποίο ήταν προβληματικό επίσης ήταν η χωρίς διακρίσεις στόχευση. Έχει ικανότητες να σημαδεύσει το Ισραήλ συγκεκριμένους τομείς, αλλά χρησιμοποίησε τη λογική των συνολικών βομβαρδισμών Κάτι το οποίο έβλαψε φυσικά και κατεδάφισε νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες, ε, τεμένη, ε, γραφεία των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Πέντε τόνοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έβρεξε πολεμοφόδια στη Γάζα στα πλαίσια της επιχείρησης του 2014. Τέσσερα παραδείγματα είναι το Μπαϊτ Χανούν, το Σεζάγια, θα σας έδειχνα και ένα φιλμ από τους βομβαρδισμούς αυτούς, αλλά δεν έχω χρόνο. Να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στο Σεζάγια ήταν εξαιρετικό. Γιατί βομβάρδιζαν για 24 ώρες συνεχώς οι Ισραηλινοί 7.000 οβίδες έπεσαν σε μια πολύ μικρή περιοχή. Ήταν τόσο εντατικός ο βομβαρδισμός που σαν στρατιωτικός ε, αναλυτής δεν μπορώ να σας δώσω μια εξήγηση ορθολογική για μια τόσο ακραία χρήση πολεμοφοδίων. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την τεχνική λογική αν θέλετε μου θυμίζει το δυτικό μέτωπο στην ε, Ευρώπη το 2018. Το 1918, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τόσο εντατικός ο βομβαρδισμός που ακόμα και οι Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είχαν ε, φρικιάσει. εφαρμόστηκε ένας μηχανισμός ο οποίος ονομάζεται Hannibal Directive. Η τακτική αυτή είναι αμφισβητήσιμη, αλλά παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να την κατανοήσουμε, γιατί ακριβώς η χρήση των πολεμοφοδίων είχε σαν στόχο το να μην απομακρυνθούν η κρατούμενοι. You will find that was utterly and absolutely indiscriminate. Houses, cars. Έτσι ώστε να αποφευθεί η απαγωγή ενός αξιωματικού. 255 ήταν τελικά οι νεκροί από την προσπάθεια αυτή. η επιθυμία του να σώσουν ουσιαστικά έναν Ισραηλινό κρατούμενο αυξάνει τον αριθμό των απολειών ε, των ε, Παλαιστινίων ακόμα και αν πρόκειται για μάχους γυναίκες και παιδιά. Θα περάσω από την άλλη πλευρά τώρα της ε, ζώνης προστασίας Ταυτόχρονα με αυτές τις ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπήρξε περιορισμός ε, της ε, περιοχής της θαλάσσιας, της ζώνης της οικονομικής της Γάζα, που περιλαμβάνει επίσης και αρκετό φυσικό αερίο το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της περιοχής αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Βλέπετε το σημείο Μάρι Β, το οποίο χρησιμοποιούν και αντλούν φυσικό αέριο μετά από τη ρύθμιση και την συμφωνία με την Αίγυπτο, ε, δεν είχαν την δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερίου και άρχισαν να χρησιμοποιούν το τοπικά διαθέσιμο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποια από αυτά τα πεδία φυσικού αερίου βρίσκονται ίσως και στα διεθνή σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα και ίσως να ανήκουν σε άλλη χώρα παρότι το χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες. Πρόσφατα ακούγεται ότι ένα κονσόρτιουμ συμφώνησε να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Αιγύπτου, Ισραήλ και Κύπρου, μέσω της Κύπρου να υπάρξει ένας αγωγός προς την Ελλάδα για την κάλυψη αναγκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πρώτη σύσταση την οποία δίδω προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακόλυθρη. Να μην υπάρξει εισαγωγή φυσικού αερίου από τη συγκεκριμένη περιοχή ή τουλάχιστον ένα τμήμα της περιοχής αυτής ε, δεν έχει πρόσβαση στον εθνικό του πλούτο. Ένας αγωγός ο οποίος θα περνά από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη προέρχεται από μια περιοχή η οποία υποφέρει, ε, είναι στο επίπεδο της καταστροφής και θα ήταν ε, ύβριστο να κάνουμε κάτι τέτοιο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τη χρήση των πυρομαχικών. Εγώ είμαι στρατιωτικός, ήμουν στρατιωτικός 42 χρόνια και αναλυτής στρατιωτικός για 20 περίπου. Είναι σαφές ότι οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο οπλικό είναι εξίσου αποτελεσματικές και μπορεί ε, πολύ πιο σκληρές από τεχνολογίες που είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιήθηκε Απεμπλουτισμένο ουράνιο. όπως επίσης ε, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ε, χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες από καουτσούκ ή ε, λάστιχο. Τεχνικά δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά η σύστασή μου είναι η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθουν λίγο στην υπόθεση αυτή, να επανεξετάσουν και να δουν τι είναι σωστό να χρησιμοποιείται και τι όχι. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αν μια σφαίρα έχει σαν στόχο το να ακυρώσει αν θέλετε μια ανθρώπινη παρουσία, τότε ακριβώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συγκεκριμένη στιγμή, αλλά όχι για όλη του τη ζωή γιατί το να τιμωρήσει κάποιον και να τον καταστήσεις άκυρο για όλη του τη ζωή σημαίνει ότι είναι μια στρατηγική επιλογή που πρέπει να καταδικαστεί. Ευχαριστώ κύριε Συνταγματάρχα. Μαχμούτ Αμπτουραχμάν του Κέντρου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Λωρίδας της Γάζας. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση της ε, αντιπρόσωπης, ε, συγγνώμη, της ε, Παλαιστίνης και Τζον, Ντέσμοντ, Έιμι με βοήθησαν πολύ για να συντάξω την παρουσίασή μου που ελπίζω να μην σας φανεί βαρετή. Είμαι μέλος ε, του Γραφείου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εδώ και 17 χρόνια και έχουμε ασχοληθεί και με ε, ζητήματα διαφορών. Για 10 λεπτά, αν μου επιτρέπετε, θα προσπαθήσω να προβάλλω το περίπλοκο επιχείρημα ότι υπάρχει άμεση ανάγκη παρέμβασης διεθνών μηχανισμών όπως αυτούς που περιέγραψε ο Τζον για ένα λόγο διότι δεν λειτουργούν οι κανονικά προβλεπόμενοι μηχανισμοί και με την άμεση συμμετοχή μας από το 2009 το έχουμε δει αυτό. Έχουμε υποβάλλει εκατοντάδες προσφυγές ασταστικά και ποινικά Ισραηλινά δικαστήρια με αποτέλεσμα σχεδόν μηδέν. Για να αρχίσω με την πιο πρόσφατη. 35 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε διαμαρτυρίες από ε, πραγματικά πειρά. Να μην επαναλάβω όλα τα νούμερα που είπατε, αλλά η πρώτη απώλεια στις 30 Μαρτίου από οβίδα πυροβολικού στην αυγή, δηλαδή στις πολύ πρωινές ώρες κατά δύο γεωργών. Ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε βαριά. Δήλωση του Ισραηλινού στρατού. Α, αυτοί οι δύο τύποι μας φάνηκαν ύποπτοι. Δρούσαν ύποπτα λοιπόν και γι' αυτό τους έριξαν μια οβίδα. Εμείς ζητήσαμε έρευνα. Αρχικός Απορρίφθηκε η προσφυγή μας, μετά όμως από διεθνή πίεση έγιναν κάποιες έρευνες, δηλαδή ανοίγει κάπου ένα παραθυράκι. Αρκεί αυτό. Εμείς νομίζουμε πως δεν αρκεί. Κάθε κράτος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έχει το καθήκον να διερευνά όταν λαμβάνει καταγγελίες ότι οι εθνικές του ένοπλες δυνάμεις έχουν ενδεχομένως ε, διαπράξει εγκλήματα είτε στη δική τους επικράτεια ή σε επικράτεια άλλης δικαιοδοσίας και εφόσον δεν το πράξει αυτό και δεν διώξει τις πράξεις αυτές αυτομάτως ξεκινά να ισχύει η αρχή της συμπληρωματικότητας όπου εμπλέκονται τότε διεθνείς μηχανισμοί. τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολους καιρούς η λόγια της Γάζας τρεις μίζονες επιθέσεις και εν τω μεταξύ σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στη ζώνη προστασίας, buffer zone δηλαδή, με πολλά θύματα, ανθρώπινες ζωές και βεβαίως και την αξιοπρέπεια του πληθυσμού. Μερικά από τα νούμερα που έχουμε από την επιχείρηση Cast LED, 1410 νεκροί, 70% άμαχοι, πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων ανθρώπων, χειρότερα από την άλλη επιχείρηση Protective Edge, όπου και εκεί είχαν πολλά θύματα. Αυτό για το οποίο εμείς παραπονούμεθα και καταγγέλουμε είναι περιπτώσεις όπου έχουμε ενδείξεις ότι έγιναν κάποια, κάποιες παραβιάσεις, παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης, της τέταρτης συνθήκης των αρχών του διεθνού δικαίου, παραβίαση της αρχής της διάκρισης, δηλαδή να στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και όχι στόχους αμάχων, αναλογικότητα και ούτω καθεξής. Αυτά λέει το διεθνές δίκαιο. Θυμούμε όμως καθαρά το 2009 ήμουν εδώ στις Βρυξέλλες και μετά πέρασα και από το Βερολίνο και είχαμε έρθει να καταγγείλουμε την συμπεριφορά του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια της επιχείρησης Cast Led και τις ποινικέ μας προσφυγές επειδή ε, ε, ευλήθησαν νοσοκομεία, άμαχοι και ούτω καθεξής. Είχαμε, είχαμε σοβαρές ενδείξεις για όλα αυτά και καταγγείλαμε τις Ισραηλινές αρχές και η απάντηση που λάβαμε ήταν το Ισραήλ δημοκρατία. Έχει πολύ προωθημένο ε, σύστημα απονομής δικαιοσύνης να πάτε να βρείτε το δίκαιο σας εκεί. Αυτό μας είπαν. Είναι προφανές ότι χρειάζεται άλλου είδους συζήτηση. Δεν αρκούν υποσχέσεις. Πολλά συνέβησαν από τότε έχουμε κάνει προσφυγές κατά της Protective Edge και επιθέσεων κατά παιδιών, παιδιά που έπαιζαν στην παραλία, κατά της στόχευσης ε, σε ε, ιδιωτικές κατοικίες, δωδεκάδες ολόκληρες, επιθέσεις κατά νοσοκομείων, βασανιστήρια, κακομεταχείριση αμάχων από στρατιωτικούς και αστυνομικούς στο Ισραήλ, καταστροφή μη στρατιωτική υποδομή, αλλά και άμεσε επιθέσει κατά καταφυγίων των Ηνωμένων Εθνών, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδε χιλιάδε αμάχων και αυτό έγινε πέντε φορέ στη διάρκεια τη ε, επιχείρηση Protective Edge. Κάναμε όπως απαιτείται από το δίκαιο, δηλαδή θεμελιώσαμε τι υποθέσει μα και στείλαμε εκατοντάδε καταγγελίε μέσω των εταίρων μα στι Ισραηλινέ αρχές το σύστημα του Ισραήλ απαιτεί οι καταγγελίε να υποβάλλονται σε ένα από δύο όργανα, είτε στην στρατιωτική εισαγγελία, και είχαν τότε ένα μηχανισμό που τον έλεγαν Fact-Finding Assessment Mechanism, και αναφέρθηκε αυτό και σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα, το κάναμε αυτό και πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια και μπορούμε να πούμε λίγα λόγια για το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί και γιατί νομίζουμε ότι δεν κάνουν τίποτα. 60% και παραπάνω από τις προσφυγές που κάναμε δεν προχώρησαν έως τώρα. Ούτε μια λέξη δεν έχουμε ακούσει για αυτές. Μόνο 2% των προσφυγών μας, των καταγγελιών μας που στείλαμε ως οργάνωση, άρχισε να γίνεται ποινική έρευνα και σε καμία απολύτως δεν έγινε συγκεκριμένη δίωξη σε κάποιον ε, στρατιωτικό. Κάποιο στρατιωτικό ε, κυνήγησαν επειδή χρησιμοποίησε μια επιστοτική κάρτα για να βγάλει λεφτά. Αυτός ο μηχανισμός fact-finding λειτουργεί με τρόπο που δεν είναι καθόλου χρήσιμος, στην ουσία κολλησιεργεί, καθυστερεί τις έρευνες κάνει συνεντεύξεις, δηλαδή παίρνει καταθέσεις μόνο από στρατιωτικούς μάρτυρες, εξετάζει απόρριτες πληροφορίες, δεν μοιράζεται μαζί μας τις πληροφορίες για το πώς καταλήγει στο εάν θα αρχίσει ποινική έρευνα ή όχι, κλείνει βιαστικά τις υποθέσεις και μιλούμε για έρευνες. Υπάρχουν όμως πρότυπα, πρότυπα, συγγνώμη, πρότυπα από το Διεθνές Εθνικό Δίκαιο για το πώς γίνονται οι έρευνε αυτέ. Πρέπει πρώτα-πρώτα να είναι άμεσε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 4 και 5 χρόνια μετά από τη χρονική στιγμή που συνέβη το γεγονό. Επίση πρέπει να είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη η έρευνα να είναι επίσης ακριβής. Αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία εξετάζουμε τις έρευνες που κάνει η εγχώρια δικαιοσύνη του Ισραήλ. Δυστυχώς αυτός ο fact-finding μηχανισμός έχει σημαντικότατα προβλήματα και σε ό,τι αφορά την ακρίβειά του και σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητά του. Είναι σοβαρότατα προβλήματα. Σκοτώθηκαν μικρά παιδιά που έπαιζαν στην παραλία και με παρουσία διεθνών δημοσιογράφων. Κάνε δεν είδε τίποτα από το στρατιωτικό προσωπικό. Ο μηχανισμός ΜΑΓ έχει λοιπόν ένα σοβαρό πρόβλημα. Στην ουσία δηλαδή έχει δύο ιδιότητες. Από τη μια συμβουλεύει το στρατό σχετικά με το ποιες επιθέσει μπορούν να κάνουν σε ποιους στόχους και από την άλλη μεριά έρχεται ο ίδιος να κρίνει εάν συγκεκριμένε επιθέσεις ήταν νόμιμες ή παράνομες. Αυτά δεν, δεν είναι χρήσιμο τελικό μηχανισμός αυτός. Και γι' αυτό κλείνει τις υποθέσεις μας βιαστικά ο μηχανισμός. Σε μια υπόθεση υπήρχε ο ισχυρισμό ότι, ακούστηκε ο ισχυρισμό δηλαδή, ότι ο Ισραηλινός στρατός στόχευσε μάχημο προσωπικό από την πλευρά των Παλαιστινίων και στην περίπτωση των Backer Boys ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα διότι ο στρατιωτικός διοικητής θεώρησε ότι τα παιδιά ήταν μαχητές της Χαμάς. Δεν έλαβε λοιπόν καμία, κανένα προληπτικό μέτρο. Απλώς στη βάση μιας υποψίας εκτόξευσαν πολλά βλήματα κατά των παιδιών και τα σκότωσαν τα περισσότερα ενώ ο στρατός έχει υποχρέωση να απόσχει από ε, χρήση όπλων εάν δεν έχει βεβαιότητα. Πρόκειται για ξεκάθαρες ενδείξεις ότι το σύστημα του Ισραηλινού στρατού δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Για τις άλλες υποθέσεις μια οικογένεια στη Ράφα όπου ο στρατός δέχτηκε ότι έκανε σφάλμα λέγοντας ότι δεν υπήρχε τελικός, όντως δεν υπήρχε θετικός στόχος μέσα στο σπίτι, ότι ήταν, είπαν, τεχνικό σφάλμα του συστήματος, έριξαν μια βόμβα στο σπίτι, τι να κάνουμε, σκοτώθηκαν, λυπούμαστε πολύ. Εμείς ζητήσαμε αποζημίωση, γιατί και αυτό έχουμε το δικαίωμα να το απαιτήσουμε από το Ισραηλινό σύστημα. σύμφωνα με το σύστημα απόδοσης ευθυνών. Και σε μια πρόσφατη υπόθεση που έχουμε, το κράτος ζητεί από το δικαστήριο να κλείσει την υπόθεση αποζημίωσης για ένα παιδί το οποίο ευλήθη στην σπονδυλική στήλη και το παιδί αυτό θα μείνει ανάπηρο για όλη τη ζωή και το κράτος είναι ανίκανο να πει αν πράγματι υπήρχε μάχημη δράση, combat action, διότι αν υπήρχε ε, combat action τότε κλείνουν το φάκελο. Τώρα λένε όμως ότι επειδή το πρόσωπο αυτό προέρχεται από τη Γάζα και θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Δεν υπάρχει λοιπόν υποχρέωση αστικής αποζημίωσης καμία υποχρέωση αποζημίωσης και για πολύ βαριά εγκλήματα. Και αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στην λωρίδα της Γάζας. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάξει και τα δικαιώματα του πληθυσμού και να τα ζυγίσει απέναντι σε ένα μηχανισμό ο οποίος δεν οδηγεί απολύτως πουθενά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Μαχμούτ. Μια στιγμή Μαρίτα, να δούμε πρώτα ποιος άλλος θέλει το λόγο. Για ερωτήσεις ή για σχολιασμό. Χάν. Μαρίτα λοιπόν. Σας ευχαριστώ όσο μιλούσατε. Θυμήθηκα τις ειδήσει που διάβασα πρόσφατα. Θα ήθελα μια αντίδραση σε αυτά. Δεν έλεγξα την αλήθεια ή όχι, πάντως ακούστηκε στις ειδήσει ότι η ρουμανική κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει την πρεσβεία της Ρουμανίας στο Ισραήλ από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Θα ήθελα να μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο, αν αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ή ελκυστικά για άλλες χώρες και πώς θα πρέπει να δράσουμε σαν βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από αυτό, έτσι ώστε να μην μπούμε σε μια κατάσταση όπου η μία χώρα μετά την άλλη θα αρχίσουν να ακολουθούν τη γραμμή του Τραμπ. Είμαι Σουηδή, είμαι σοσιαλδημοκράτης και ανησυχώ που μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση μάλιστα στη Ρουμανία το αποφάσισε. Ίσως να μην είναι και αληθές όμως. Έχετε κάποιο σχόλιο γύρω από αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, για πολύ ενημερωτικές πληροφορίες και τεχνικές επίσης λεπτομέρειες. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικά αυτά όλα για μένα. Θα ήθελα επίσης να σταθώ στην παρουσίασή σας κύριε Τζουγκάρντ. Δεν θα μπορέσω να ακούσω όλες τις απαντήσεις γιατί δυστυχώς πετάω σύντομα. Αλλά η συζήτηση αυτή που γίνεται είναι ιδιαίτερα εύθετη. Περάσαμε ένα ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα και απογοητεύτηκα από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, όχι παρόντες, που ήθελαν το ψήφισμα αυτό να έχει σαν βασικό θέμα το Χαμάς. Το θέμα αυτών που πέθαιναν στα σύνορα το συνέδεαν με το Χαμάς. Ενώ εγώ νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό είχε σαν στόχο την καταγγελία των απαράδεκτων ενεργειών που οδήγησαν στους θανάτους των νέων αυτών ανθρώπων. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν γύρω από αυτό. Η επίπτωση του Χαμάς, της ύπαρξης του Χαμάς σε σχέση με τα επεισόδια είναι σαφής. Εσείς γνωρίζετε την κατάσταση. Υπήρξε κάποια δικαιολογία Η στάση του Χαμάς ε, που δουλεύει κατά τα άλλα στην περιοχή είναι ε, ε, λανθασμένη, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Και ένα τελευταίο σημείο. Μιλήσατε για τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είναι εφόσον παραμείνουν σιωπηλές συνένοχες. Και η μετακίνηση της πρεσβείας των ΙΠΑ στην Ιερουσαλήμ είναι κάτι που δεν προκάλεσε τις αντιδράσεις που περιμέναμε. Στην ουσία δηλαδή εμείς ακολουθούμε την πολιτική του Twitter του Τραμπ. Και ο, η δολοφονία των ασθενών στα νοσοκομεία, η καταστροφή των, νοσοκομείων δεν πνίγουν την κατάσταση, τη δημιουργούν ιδιαίτερα πνιγυρή και δεν φαίνεται να έρχεται κοντά η λύση των δύο κρατών. Ευχαριστώ συνάδελφε Κάνη, ήμουν συνεισηγητή στο ψήφισμα αυτό και εκεί ήταν και η βασική μου αντίρρηση σε σχέση με το Χαμάς. Αναφέρεται επτά φορές το ψήφισμα. Και γι' αυτό ακριβώς το τέλος σωτήρισα στάση αποχής και το επεξήγησα με την ψήφο μου. Εντουάρ Μαρτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση αλλά πρώτα κάποια σχόλια. Να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο δυστυχώς για μια ακόμη φορά την μειωστή φορά 12 χρόνια μετά από την αρχή του αποκλεισμού της Λωρίδας. Ο κατάλογος των εγκλημάτων πολέμου, της καταστροφής, της δολοφονίας μεγενθύνεται. 12 χρόνια τουλάχιστον και η Ευρώπη απλά παρακολουθεί, κοιτάει αλλού. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Εμείς θα πρέπει, ε, ε, αν πούμε ότι η Ευρώπη είναι ζώο, τι ζώο θα ήτανε. εγώ θα έλεγα ότι είναι αγελάδα, γιατί οι αγελάδες βλέπουν τα τρένα να περνούν. Ωραία αγελάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για τη Γάζα. Λοιπόν, αστείο αυτό, αλλά αυτό που πρέπει να καταγγείλουμε πρώτα είναι η λεγόμενη συλλογική μας υποκρισία. Και έρχομαι εδώ και στη συζήτηση για το ψήφισμα της προηγούμενης εβδομάδας για τη Γάζα. Υπερψήφισα εγώ, γιατί είπαμε ότι ήταν καλύτερα από το τίποτα. Δυστυχώς έτσι λέμε. Καλύτερα από το τίποτα. Αλλά τώρα το καλύτερα και το τίποτα πολλές φορές είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο την υποκρισία των κρατών μας και της Ευρώπης. Παρατήρησα αυτά που είπατε επίσης ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να διωχθούν και για συνενοχή σε, εγκλήματα, σε τέλεση εγκλημάτων πολέμου γιατί δεν διευκολύνουν την δραστηριότητα του διεθνούς ποινικού ε, νομίζω λοιπόν ότι και σε νομικό επίπεδο να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί σε πολιτικό επίπεδο δεν γίνεται τίποτα. Η Ευρώπη θέλει να είναι φίλη όλου του κόσμου, και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, αλλά οι, Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνοι οι φίλοι κατάλαβαν ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι και φίλο τους, είναι μια ομάδα υποκριτών. Και αναφερθήκατε σε κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές που θα έκαναν το ίδιο λάθος να μεταφέρουν δηλαδή την πρεσβεία του στο από το Τελαβίβα. Ε, θα ήθελα να πω ότι οι μάσκες ε, πέφτουν τελικά. Και έχω την αίσθηση ότι η Παλαιστίνη και το Παλαιστινιακό δεν απασχολεί όπως θα έπρεπε πια τη διεθνή κοινότητα και γι' αυτό έστω και σε νομικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Και εδώ στρέφομαι τώρα στην κυρία Σάλαν που ασχολείται με τα ιατρικά θέματα και εγώ ε, συνεργάζομαι με την ε, οργάνωση Palm Ed που είναι μια οργάνωση Παλαιστίνιων γιατρών οι οποίοι ήρθαν να μας συναντήσουν έτσι ώστε να μας ζητήσουν βοήθεια για να ε, δημιουργήσουν μια μονάδα παραγωγής από ηλιακή ενέργεια. Ε, το πρόβλημά μας είναι ότι για να μπορέσουμε να βάλουμε τα υλικά αυτά στη Γάζα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε γι' αυτό. Κάνω δύο ερωτήσεις σύντομες. Η πρώτη είναι στην κυρία Ματέρη. Ε, είπατε για την οικονομική ε, αρρωγή. Ε, μετά την απόφαση της ζήτησης Τραμπ τον είπα για μείωση τη αρρωγή προ την Ούνδρα, έγινε μια διεθνή σύνοδο στη Ρώμη για δωρητέ πριν από λίγο καιρό. Και επειδή σε παλιότερη συζήτηση μα στην αντιπροσωπεία με Παρσίνη αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο τη Ούνδρα στη Γάζα, τον οποίο είχαμε απευθεία από εκεί, ότι για την ε, συμβολή στην παροχή τροφίμων ε, στον πληθυσμό στη Γάζα τα λεφτά αρκούν μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω τι μέτρα παίρνουμε γιατί ενδεχομένως να έχουμε μια μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία και κρίση μετά από αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και το άλλο ερώτημα μου είναι στον καθηγητή, στον κύριο Ντουκάρτ. Ανεβευθήκεται για τις αποζημιώσεις ε, που πρέπει να διεκδικήσουν από το Ισραήλ. Είναι ένα θέμα που συζητούμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Διότι όντω ε, ε, υπάρχουν καταστροφές υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω ένα παράδειγμα που δεν αφορά τη Γάζα. Τώρα θα καταστρέψουν ένα ε, σχολείο στην περιοχή των Βεδουίνων στο Καναλάχα, το οποίο έγινε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα έχουν πάρει απόφαση μάλιστα πρόσφατα από το δικαστήριο μετά από δική μα παρέμβαση και επίσκεψη τη αντιπροσωπεία μα ανεβλήθηκε αλλά υπάρχει απόφαση να καταστραφεί. Και ήθελα λίγο αυτό να μα το εξηγήσετε, δηλαδή οι διαδικασίε που πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει για να διεκδικήσει αποζημιώσει από το Ισραήλ, εκεί που καταστρέφονται με τι ε, επιδρομέ του Ισραήλ υποδομέ που ανεγέρθηκαν με χρηματοδότηση τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> και τώρα ο λόγο ε, ξεκινώ για σχόλια σύντομα από όλου. Να ξεκινήσω από τον ε, καθηγητή των προφέσεων ε, Α, sorry, ε, just... Yes, Soraya. You want, yeah. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, πρώτα η Σωράγια να ρωτήσει κάτι ακόμα. Λυπούμε, λυπούμε πολύ. Είχα άλλη συνάντηση και δεν πρόλαβα να έρθω από την αρχή και να ακούσω τι ομιλίε σα. Λυπούμε πολύ γι' αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, διεθνή κοινότητα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Τώρα με την κατάσταση Ισραήλ-Παλαιστίνης και όχι μόνο εκεί βέβαια, αλλά και αλλού βεβαίω Συρία, Ιράν και άλλα ε, μέρη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πιο ενεργό ρόλο για να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων. Εγώ πήγα πριν από ένα μήνα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη Ήμασταν μια προοδευτική αντιπροσωπεία σοσιαλιστών και δημοκρατών. Δεν μας επέτρεψαν να πάμε στη Γάζα από το Ισραήλ. Αλλά πήγαμε τουλάχιστον στην Ευρών, στη Γαμάλα, πήγαμε σε ε, καταβλισμούς Βεδουίνων και είδαμε και τις δυο πλευρές, εκπροσώπους και των δυο πλευρών. Αυτό πάντως που είδα είναι το καθεστώς apartheid, τουλάχιστον στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κάτι το τρομακτικό, διότι όταν πυροβολούν διαδηλωτέ. Μόνο επειδή διαδηλώνουν. Δεν καταλαβαίνεις πια πώς η κυβέρνηση που ό,τι θεωρώ ακροδεξιά, πώς αντιμετωπίζει τέλος πάντων την κατάσταση, την ειρηνευτική συμφωνία, το ενδεχόμενο της λύσης των δύο κρατών δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και αναφέρονται στην κατάσταση ασφάλειας, όλο λένε για κατάσταση ασφάλειας, και από την άλλη μεριά αρπάζουν όλο και περισσότερα εδάφη. Αυτά δίνουν ένα μήνυμα. Από τη δική σας γνώση τώρα και από τις εμπειρίες σας, να μας τα πείτε ειλικρινά. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε. Ποια είναι η ευθύνη μας. Εγώ ξέρω, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα από τους ειδικού. Διότι καθώς ήμουν εκεί, στη Ραμάλα και στην Ευρών, είδαμε την απογοήτευση. Και από τις δυο πλευρές. Και επίσης δεν έχουν καθόλου ε, θετικές προοπτικές για το μέλλον. Δεν ήταν καθόλου θετική. Ε, ε, θεωρώ ότι πρόκειται για μεγάλη απογοήτευση. Κάποιοι έχουν κάποιες ελπίδες, και μιλούν και για τη λύση των δύο κρατών, αλλά δεν έχουν λύσει για το πώς θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ αποκαρδιωτικό το ταξίδι αυτό. Ακόμα χειρότερο από ό,τι το περίμενα. Άρα, ξαναρωτώ, τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι, αν δεν μπορούμε να λύσουμε την κατάσταση αυτή στο προσεχές μέλλον, νομίζω ότι η σύγκρουση αυτή θα συνεχίσει να κλιμακώνεται και θα συμπαρασύρει όλη την περιοχή γιατί βλέπω εμπλοκή και στις συζητήσεις βλέπω ε, να εμπλέκεται στις συζητήσεις και φόβος το τι μπορεί να γίνει με το Ιράν, ο πόλεμος στη Συρία, οι χώρες του Περσικού. Είναι ένα μεγάλο ανακάτεμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ Ο καθηγητής Ντουγκάρντ. Δεν νομίζω ότι απευθύνατε όλες τι ερωτήσει σα σε μένα. Πρώτα για τη Ρουμανία. Διάβασα και εγώ την είδηση ότι σκέπτονται οι Ρουμάνοι να μεταφέρουν την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Εδώ χρειάζεται να το ψάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ως σώμα, ως ενότητα ξεκαθαρίσει ότι, πρόκειται, ότι είναι κάτι το αντίθετο στην πολιτική προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων να μεταφέρουν την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Γιατί έμεσα δείχνουν έτσι έγκριση των πρακτικών του Ισραήλ. Η άλλη ερώτηση σας, η πιο τελευταία, ήταν πολύ σημαντική. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση αυτή. Το πρώτο είναι να σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Να σταματήσει να συνεργάζεται με το Ισραήλ. Εγώ είμαι Νότιο Αφρικανό, Οι Νότιο Αφρικανοί υπέστησαν παντός είδου κυρώσει από οικονομικές μέχρι στον αθλητισμό. Το Ισραήλ προχωρά σε μια πρακτική που είναι πολύ παρόμοια. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ πρόσφατα ομάδες και, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται το Ισραήλ να συνεργαστεί μαζί τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι καθαρό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει το Ισραήλ και συνεργάζεται μαζί του. τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, αυτό που πρέπει να αναμένει κανείς είναι να σταματήσει η συνεργασία αυτή. Και αυτό θα έχει και σημαντική επίπτωση. Το ίδιο για τις ε, απαιτήσει αποζημίωσης. Εάν το Ισραήλ καταστρέψει μια υποδομή την οποία έχει πληρώσει μια κυβέρνηση μιας χώρας, αυτή η χώρα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Έχω ακούσει και στο Βελίκη στην Ολλανδία ότι σκέπτονται κάτι τέτοιο, αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένη ανάληψη δράση κατά του Ισραήλ όταν καταστρέφει υποδομές. Αλλά πρέπει πρώτα-πρώτα η στενή συνεργασία μεταξύ Ένωση και Ισραήλ να σταματήσει. to be short. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Πρώτα η κυρία Ματέρη. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που θέσατε το ζήτημα της ε, χρηματοδοτικής κρίσης της Ούνρα. Αρχές του χρόνου ακούσαμε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών που για πολλά χρόνια ήταν σημαντικός και σταθερός δωρητής της Άνωρα. Είπε λοιπόν ότι διακόπτει τη χρηματοδότηση με 300 από τα 364 εκατομμύρια δολάρια μας αφήνει με ένα τεράστιο έλλειμμα. 246 εκατομμύρια. Τεράστιο κενό. Στις 15 Μαρτίου έγινε διάσκεψη δωρητών στη Ρώμη με συμμετοχή 75 αντιπροσωπιών και με σημαντική στήριξη προς τον οργανισμό μας από κάθε άποψη και δεσμεύτηκαν να καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια. Τα μισά από αυτά το Κατάρ και τα άλλα μισά από πάρα πολλέ χώρε όλου του κόσμου. Είμαστε ευγνώμονε στη διεθνή κοινότητα για την έκφραση αυτή αλληλεγγύη η οποία ενισχύει την εντολή μα και ταυτόχρονα και οι περαιτέρω υποσχέσεις που δόθηκαν κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αναφέρω τις πιο σημαντικές δωρεές, έτσι είναι, της ε, βεβαίως παραμένει ένα κενό ιδίω για τη διανομή τροφίμων μπορεί αυτή να υποστεί ζημία και να μην μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τον έκτο μήνα του 2018 και το πρόγραμμα παροχής εκπαίδευσης εφίσταται βλάβη. Έχουμε 267 σχολεία με 270.000 παιδιά Παλαιστινίων προσφύγων. Θα ολοκληρώσουν το σχολικό έτος τον Ιούνιο, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα, μπορέσει, θα μπορέσουν όλα αυτά τα σχολεία να ξανανοίξουν το τέλος Αυγούστου. Ο εκπρόσωπος μας Βρυξέλλε τόνισε ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, διότι 270.000 παιδιά έξω από το σχολείο κανένας δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει στη Γάζα και από την άποψη της ασφάλειας και σταθερότητας της κατάστασης. Μπαίνει όμως το ερώτημα πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και υπό ποια σημαία, εάν δεν είναι η σημαία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που καταθέτουμε απέναντί σας ως Ευρωβουλευτές και είναι πραγματικά βαριές και σοβαρές απειλές που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Τι μπορεί να γίνει η σύνθεση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν δείχνουν πόσο σοβαρές είναι οι προσπάθειες που κάνουμε να διευρύνουμε την βάση δωρητών. Έχουμε την ισχυρότερη βεβαίω βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είμαστε πραγματικά ευγνώμονε. Επίση από χώρε του Περσικού, την Ινδία και αλλού, από όλε τι πλευρέ, από όλε τι γωνιέ του κόσμου για την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, παρακαλούμε να συνεχίσει να μας υποστηρίζει και να αυξήσει την υποστήριξη και στο χρηματοδοτικό επίπεδο και στο πολιτικό, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού μέσω πρόθεσμα. Αυτό το εκτιμούμε πολύ, εν ώψη βεβαίως και της ψήφισης του επόμενου προϋπολογισμού που η σύνταξή του έχει αρχίσει. Και τέλος, επειδή ο κ. Καν έφυγε και ζητούσε να μάθει για τις διαδηλώσεις, Αυτά τα είπαν και άλλοι εδώ του πάνελ. Εμεί θεωρούμε ότι παρόλο μπορεί να συμμετέχουν κάποιοι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες με δικές τους ατζέντε και με δικά τους συμφέροντα, ο μεγάλος αριθμός των διαδηλωτών φαίνεται να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους με ειρηνικό τρόπο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω την σημασία του να είναι εγγυημένο το δικαίωμα των διαδηλωτών αυτών να διαδηλώνουν ειρηνικά και να προστατευτούν οι πρόσφυγες στην Λωρίδα της Γάζας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω αυτά τα οποία ακούστηκαν ήδη. Στα πλαίσια της εμπειρίας μας, η κοινωνία των πολιτών είναι αυτή η οποία ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Υπάρχουν πέντε στρατόπεδα στην συνοριακή περιοχή, στις οποίες διεξάγονται ε, εκπαιδευτικές διαδικασίες, ε, οργανώσεις ε, συμβάντων, εορτές κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές ειρηνικές διαδικασίες ε, που εντάσσονται όλα στις διαμαρτυρίες αυτές. Τώρα για τα 12 χρόνια που η Ευρώπη είναι ένας απλός παρατηρητής. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ε, να πούμε επίσης ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι εφαρμόζονται το διεθνές δίκαιο στη δική τους περίπτωση. Παρόλα αυτά θέλουν να συνεχίζει να εφαρμόζεται και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι πραγματικοί άνθρωποι, δεν είναι ψεύτικα ομοιώματα ανθρώπων, έχουν δικαιώματα και πρέπει τα δικαιώματα αυτά να γίνουν σεβαστά. Νομίζω πρέπει να υπάρξει τέλος στην ατιμορρησία. Αναφερθήκατε επίσης και στη συνάντηση με την οργάνωση των Παλαιστινίων ε, Ιατρών, το PALMAID. Είναι σημαντικά για τους ε, ιατρούς, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες ειδικότητε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με την κάλυψη των ηλιακών ε, μορφής, μάλλον μηχανημάτων παραγωγής από ηλιακή ενέργεια ηλεκτρισμού. Ε, υπάρχει μια τρομακτική κρίση ηλεκτρισμού στην Γάζα. Πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους, αλλά ε, από ό,τι φαίνεται λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να αναλυφθεί βασικά ε, ξεκάθαρη δράση έτσι ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός. Δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο στις καταγγελίες, αλλά να αναλυφθεί δράση για την απόδοση ευθυνών. Είναι δύσκολο για τον κόσμο να καταλάβει ποια είναι η κατάσταση επιτόπου. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση, είναι ιδιαίτερα σύνθετο το σύστημα ελέγχου των Παλαιστινίων, αλλά γενικά απλά μπορούμε να πούμε ότι ζουν μια αδικία και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και αυτό το θέμα το συζήτησα με Παλαιστίνιους γιατρούς και εγώ και θα ήταν μια καλή ιδέα να προωθήσουμε την ηλιακή ενέργεια για τα νοσοκομεία γενικότερα στη Λωρίδα της Γάζας χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταγματάρχης Τρέιβες. It's not working? Working. question of Hamas and terrorism. Um, ε, σχετικά τώρα με το Χαμάς και την τρομοκρατία. Το πραγματικό πρόβλημα με αυτού του είδους την τρομοκρατία είναι η χωρίς διακρίσεις πυροβολισμη στο εσωτερικό μιας ελεύθερης κατά τα άλλα υποτίθεται χώρας. Εδώ πρέπει να κάνουμε κριτική στην κατάσταση, πρέπει να καταδικάσουμε την κατάσταση. Το 2010 στην αποστολή έρευνας που είχαμε κάνει καταδικάσαμε τη συμπεριφορά του Χαμάς. Καταλαβαίνετε ότι η τρομοκρατία θα μπορούσε να τεκμηριωθεί. Ξέρετε τι συνέβη στην Ιρλανδία σαν παράδειγμα αλλά παρόλα αυτά οι τρομοκράτες θα πρέπει υποτίθεται να πράττουν με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει τους αμάχους πριν από οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω ζούσα στο Ισραήλ σε μια περιοχή που βομβαρδίζεται τακνικά με ε, πυράβλους κατιούς από το Λίβανο και υπάρχει μάλιστα και ένα μέλος της οικογένειάς μου εδώ που γνωρίζει πόσο πραγματικά άβολη ήταν αυτή η κατάσταση. Βέβαια τα θύματα ήταν ε, μηδενικός ο αριθμός τους, αλλά παρόλα αυτά ήταν τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργούσαν οι βομβαρδισμοί και η ψυχολογική πίεση. Εμείς λοιπόν στην αποστολή έρευνας που κάναμε εντυπωσιαστήκαμε με τους Ισραηλινούς πολίτες και στο Αμάν και στη Γενέβη που είχαν πει ότι επηρεάζονται και από τις σιρήνες και από τα σχολεία τα οποία οδηγούν τα παιδιά σε καταφύγια αλλά τους έκανε εντύπωση επίσης και η απουσία οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου σε περιοχές που εξετίθετο σε κίνδυνο. Λοιπόν, τώρα η περιοχή αυτή, η ενδιάμεση περιοχή προστασίας είναι, όπως σας είπα, η περιοχή στην οποία υπάρχουν τα περισσότερα θύματα σε αιτήσια βάση. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία να καταδικάζουμε το Χαμάς για τις ροκέτες που, με τις οποίες βομβαρδίζει το Ισραήλ και να μην μιλάμε για τους πυροβολισμούς του Ισραήλ προς το εσωτερικό της Λωρίδας. Λοιπόν, ή το ένα ή το άλλο. Ευχαριστώ. Ο Μαχμούντ έχει το λόγο. Θα πρέπει να είσαι σύντομος, Μαχμούντ. Για το θέμα του Χαμάς πάλι, να πω ότι υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για τους οποίους δεν ερωτεύεται κανείς το Χαμάς εισαγωγικά. Πολλοί από τους λόγους αυτούς έχει να κάνει και με τη μεταχείριση του πληθυσμού ε, από την ηγεσία στη Γάζα και ασκούμε κριτική σε αυτό το οποίο καθημερινά κάνουμε. Αλλά το ότι το Χαμάς προετοίμασε τις διαδηλώσεις, το ότι το Χαμάς χρησιμοποιεί σαν τείχος προστασίας τους διαδηλωτές ε, έτσι ώστε να μετακινεί τους πληθυσμούς με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι μαχητές του. Ε, όχι βέβαια, δεν ισχύει αυτό, το διερευνήσαμε και δεν ισχύει. Το να δικαιολογεί κανείς τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων και να κατηγορεί στην συνέχεια το Χαμάς ε, είναι απαράδεκτη. και πριν από την πρώτη Παρασκευή της επίθεσης ε, οι δηλώσεις ε, της κυρίας Μογκερίνη και της γερμανικής κυβέρνησης ε, που συμφώνησε με αυτές τις λογικές της Ισραηλής κυβέρνησης είναι απαράδεκτες. Περιμένουμε το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αντικειμενικό, να είναι τεκμηριωμένο και να μην βασίζεται σε φημολογίες οι οποίες είναι πληρέστατα ανεπιβεβαιωτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε καμία περίπτωση μέχρι τώρα. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνουν από εδώ και πέρα. Είπαμε ότι η απόδοση ευθυνών είναι το σημαντικό. Ε, πρέπει να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. έχει ξεκινήσει η διαδικασία εισόδου της Παλαιστίνης στο διεθνές ποινικό. Θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ένταξη της Παλαιστίνης. Τώρα, ε, θα πρέπει να δούμε ότι πέρα από την κατάσταση στα Ιεροσόλυμα, η κατάσταση στη Γάζα είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όπως είναι πρέπει να αμφισβητηθεί αμέσως η κατάσταση στη Γάζα και ο αποκλεισμό, γιατί αλλιώς η Γάζα πράγματι ε, θα χαθεί, μια ολόκληρη γενιά θα χαθεί. Συνεπώς όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν μέσω ε, της ε, τήρησης των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απλά σε επίπεδο σεβασμού διεθνούς δικαίου, όχι σε επίπεδο πολιτικής. Πριν να δώσω τον λόγο στον ε, ε, πρόεδρο της ε, ΤΡΟΑ, τον συνάδελφο Παντζέρη, ήθελα να σχολιάσω δύο πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του delegation όλους τους ομιλητές. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που είπε η Σωράγια ε, μου έτυχε να επισκεφθώ πολλές φορές την Παλαιστίνη. Take I Επισκέφθηκα πολλέ φορέ την Παλαιστίνη και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο ένα και περισσότερο νιώθει αυτό που λέγεται για το Apartheid. Και το χειρότερο είναι ότι χωρίζουν του Παλαιστίνιου. Οι Παλαιστίνοι είναι σε διάφορε ομάδε. Είναι διαφορετική η ζωή των Παλαιστινίων στη Ραμάλα, διαφορετική στη Βιθλέμ, διαφορετική στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ε, με διαφορετικά προβλήματα οι Άραβες, Παλαιστίνοι, οι πολίτε του Ισραήλ. Ε, αυτό μου θυμίζει ε, περισσότερο, ε, δεν πήγα ποτέ στην Νότια Αφρική καθηγητή, έχω διαβάσει πολλά για την Νότια Αφρική, αλλά μου θυμίζει αυτό τα πάντουσταν στην Νότια Αφρική και πώς διαχωρίζουν όλους τους πολίτες και ασκούν πίεση. Βεβαίω η χειρότερη κατάσταση είναι στη Γάζα. Και είναι ένα θέμα, επειδή το ανέφερε η Σωράγια, ένα θέμα που πρέπει να ασκήσουμε πιέσει και ω Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πατρική Εκπρόσωπο δεν είναι παραδεκτό, είναι ανεπίπτωτο θα έλεγα να μην επιτρέπεται η επίσκεψη Ευρωβουλευτών στην Λωρίδα της Γάζας. Δοκίμασαμε πολλέ φορέ και σαν επίσημη αντιπροσωπεία δεν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ο μόνο που είχε τη δυνατότητα για μερικέ ώρε πέρσι ήταν ο πρόεδρο τη επιτροπή Πάτζετ. Ε, πολύ περισσότερο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτά έργα, συμμετέχει στη στήριξη τη ανθρωπιστική βοήθεια και το θεωρούμε απαραδεκτό. Και το τελευταίο να πω ότι επειδή γίνεται πολλέ αναφορέ για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ, γίνεται συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και είμαι ένα από αυτού που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μια πίεση για να δούμε πώ υλοποιείται η Συμφωνία Σύνδεση και κατά πόσο αυτή η Συμφωνία Σύνδεση πρέπει να απαγοποιηθεί. Από τη στιγμή που το Ισραήλ παραβιάζει κατάφορα το άρθρο 2 που αναφέρεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άρθρου 2 αυτή τη συμφωνία σύνδεση. Και ε, πέρα από αυτά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα ε, και να διαβεβαιώσουμε την εκπρόσωπο τη Ούντρα ότι πρέπει να στηρίξουμε την Ούντρα. Η Ούντρα επιτελεί έναν σημαντικό ανθρωπιστικό ε, ρόλο και στόχο για όλους τους Παλαιστίνους και ιδιαίτερα στη Γάζα, στην οποία χωρίς την υποστήριξη τη Ούντρα δεν μπορεί να επιβιώσει ο κόσμο στη Γάζα. Ευχαριστώ για την παρουσία όλων. Ο λόγο τώρα στον ε, κύριο Μπατζέρη για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Bene, grazie, grazie a tutti. Io brevissime considerazioni Πρέπει eh, eh, να διευκρινίσω ότι ήδη σχετικά με την ε, μεταφορά της ε, πρεσβείας της Ρουμανίας ε, στην Ιερουσαλήμ είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε ακόμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί, όχι μόνο γιατί δεν συμφωνούμε, γιατί έρχεται σε αντίφαση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως είπε η ύπατη εκπρόσωπος πάνω σε ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει να σεβαστούμε ε, τις διαφορετικές απόψεις και να δούμε τι ακριβώς επιθυμεί η ρουμανική κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό θέμα, ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής περισσότερο. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Παλαιστίνη, το Παλαιστινιακό, δεν είναι πια ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο στο παρελθόν. Και το Ισραήλ μέσα από το χρόνο προσπαθεί να αποτρέψει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους όχι μόνο μέσω της απικιοποίησης, αλλά μέσω και της χρήσης της γάζα σαν μοχλοπίεσης. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα εδώ. Στις εσωτερικές συγκρούσεις προστίθεται και το διεθνές ε, πρόβλημα της ε, αντιπαράθεσης Κατάρ Σαουδικής Αραβίας. Είναι σημαντικό για την περιοχή, είναι σημαντικός χρηματοδότης ε, της Λωρίδας της Γάζα το Κατάρ και η σύγκρουση αυτή έχει συνέπειες. Πρέπει επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η Ευρώπη είναι από τους βασικούς δωρητές οικονομικής βοήθειας της περιοχής και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Αν τώρα η ανθρωπιστική, κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε να ελαφρυνθεί, η Ευρώπη θα συνεχίσει να κάνει αυτή την προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ε, πρωταγωνιστής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την υπόθεση αυτή. Μια τρίτη σκέψη Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί η κατάσταση της ζωής των Παλαιστινίων είναι εξαιρετικά άσχημη και συνέπεια άμεση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από το Ισραήλ. Και είναι σαφές ότι ε, έχουμε, έχουν καταστραφεί όλοι οι παράμετροι οικονομικοί και κοινωνικοί στη λωρίδα της ε, Γάζα και στην ουσία δεν θα μπορεί να επιβεβαιώσει η περιοχή αυτή μετά το 2020. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει επιτέλους αυτός ο αποκλεισμό. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική δράση για να αλλάξει η πολιτική του Ισραήλ. Και τέλος μετά από τα τελευταία επεισόδια Νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα ε, σαφώς θα πρέπει να δώσει εγγυήσεις έτσι ώστε να υπάρξει απόδοση ευθυνών μέσα από μία αντικειμενική ε, έρευνα. Νομίζω ότι το θέμα της ατιμορρησίας είναι ένα βασικό πρόβλημα για την κατάσταση σήμερα στην περιοχή και αν δεν ε, αντιμετωπιστεί θα συνεχώς θα χειροτερεύει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν υπογραμμίσει το πώς έχει η κατάσταση και έχουμε υπογραμμίσει το τι είναι απαραίτητο να γίνει από εδώ και πέρα. Αγαπητές συμπρόεδρε, θα πρέπει λοιπόν στο τέλος αυτής της συνάντηση να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα μικρό κείμενο, κοινό κείμενο, το οποίο να στείλουμε σε όλους τους συναδέλφους μας λέγοντας ότι ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να πρωταγωνιστήσει ακόμα περισσότερο στην υπόθεση αυτή και να προσπαθήσει να επηρεάσει τον ρόλο τον οποίο παίζει το Ισραήλ. Αυτά.